Meine Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, δεν είναι ακόμα παρόντες πολλοί συνάδελφοι. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας πω ότι έχουμε τις εξής τροποποιήσεις. Το σημείο 5 θα ξεκινήσουμε από το σημείο 5. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Το σημείο 8 είναι η Καλιφόρνια, το σημείο 7 θα είναι η κυρία Τσαβέλα, το σημείο 6 η έκθεση Beauty Coffer και το σημείο 9 η συνεδρία των συντονιστών. Το σημείο 4 αναβάλλεται μέχρι αύριο. Μία παράκληση παρακαλώ Ε, η ημερήσια διάταξη εκπονείται από τη γραμματεία, γραμματεία πολύ νωρί. Βέβαια δεν είναι αρκετή εδώ πέρα για να το ανακοινώσω, αλλά δεν μπορούμε συνέχεια ε, να τροποποιούμε την ημερήσια διάταξη επειδή κάποιο δεν μπορεί τελευταία στιγμή. Πάντα τελευταία στιγμή κάποιο παίρνει τηλέφωνο και λέει ότι δεν μπορώ στι 12 πρέπει να φύγω, στις 5, από τι 5 και μετά δεν θα είμαι. Ε, δεν, δεν λειτουργεί όμω το θέμα έτσι. Σα παρακαλώ λοιπόν να μην γίνονται τροποποιήσει στην ημερησία διάταξη και μία παρατήρηση, ε, μία ανακοίνωση του Προέδρου. Είχαμε μακρά συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και την ε, Ήτρε. Δυστυχώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε κάποια θέματα ε, για την ε, έκθεση αυτή έχει ε, ψηφίσει για θέματα όπου είχαμε εμεί την αρμοδιότητα. Έχω διαμαρτυρηθεί στην διάσκεψη προέδρου, των Προέδρων θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια, πρέπει να αναβληθεί, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες ε, της Ολομέλειας ε, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Εγώ θα το αναφέρω στη μικρή Ολομέλεια, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να δεχτούμε τους κανόνες αυτούς ε, και η εισηγήτρια... Τουλάχιστον για τα δύο σημεία όπου ε, παραβιάζεται η αρμοδιότητά μας, ε, θα υποβάλουμε ε, απευθείας τις τροπολογίες μας στην Ολομέλεια ως τροπολογίες Επιτροπής. Αυτό είναι το μόνο που, να, που μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζω να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 5. Μπορεί κάποιο να με ενημερώσει αν είναι ενημερωμένοι όλοι οι, οι, Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Ε, αυτό θα είναι το σημείο 4 στη μερίσια διάταξη. Η Λένα Εκ είναι αρμόδια, δεν είναι όμως εδώ η συντηρητήρια της νομοδότησης. Δεν ξέρω αν είναι εδώ οι άλλοι συγητές. Πάρα πολύ ωραία, τι να πω. Κάναμε τι ανακοινώσει του Προέδρου. Να, να ψηφίσουμε μία φορά, πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι θα μάθει ο κόσμος. Θα ich noch Έχω μια εναλλακτική πρόταση. Ε, αλλά ούτε και αυτή μπορώ να την εφαρμόσω, διότι δεν είναι εδώ η αντιπρόεδρο που έχει γενέθλια, θα μπορούσαμε να τη τραγουδήσουμε όλη χρόνια πολλά. Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann es machen. Θα μπορούσα, δεν είναι καλό βέβαια αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να πάμε στο σημείο 8 που έχουμε την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπεία τη Ήτρες στην Καλιφόρνια. Ε, δεν είναι όμω ε, κανένα από εδώ που θα συμμετάσχει στο ταξίδι, αλλά έτσι δεν μπορεί και κανένα να μου φέρει αντίρρηση. να το κάνουμε αυτό, να μεταφέρουμε αυτό. Καλά, δεν έχει πολύ σημασία. Στο κάτω-κάτω συμφωνούμε. Πάντως ήταν ε, εξαιρετικό το ταξίδι αυτό. Ζητήσαμε ταξίδι στην ε, Καλιφόρνια ε, ε, για να ασχοληθούμε με την καινοτομία, να δούμε τι εμπειρίες έχουν εκεί. Είχαμε μια μεγάλη αποστολή, παρότι φύγαμε με με πολύ μικρή προειδοποίηση, ήταν όμως εξαιρετική η προετοιμασία και έχει υποβληθεί έκθεση στην ε, Επιτροπή των Προέδρων των Αποστολών. Θέλαμε για κάποια σημεία που μας ενδιαφέραν ιδιαίτερα, ε, θέλαμε να συζητήσουμε περισσότερο και Κάποιοι από τους ε, συναδέρφους ε, θέλαμε να τονίσουμε ε, κάποια θέματα. Ο συνάδελφος Μπίτι Κόφερ πρότεινε να έχουμε μία μέρα γεφυρώματος Ευρώπης-Καλιφόρνιας. αυτό όμως δεν πέτυχε και θέλαμε να ρωτήσουμε τη σχετική διεύθυνση γιατί ε, απέτυχε αυτό και θέλαμε να επαναλάβουμε την πρόταση αυτή. Δεύτερον, θέλαμε να, έχουμε, να υποβάλουμε ερώτημα προς την Κομισιόν ως Επιτροπή ρωτώντας τι μηχανισμοί συνεργασίας υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Καλιφόρνια, διότι ακούσαμε τόσες εντυπωσιακές ιστορίες, θα θέλαμε πολύ να δούμε αν υπάρχουν Συνεργασίε ανάμεσα ε, με την Κομισιόν ή με το Κοινοβούλιο και εάν ναι ποιες. Ε, τρίτον, ενδιαφέρον ήταν το θέμα ε, της ρύθμισης σε περίπτωση Ε, Είδαμε κάποιους που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στην Καλιφόρνια μας εξήγησαν πόσο δραματική είναι η κατάσταση σε περίπτωση αφαιρεγκαιότητα ε, και το πρώτο βήμα στην ε, περίπτωση αυτή θα ήταν να καταβάλουμε προσπάθειες να μάθουμε από την Κομισιόν τι αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρώπης ε, όσον αφορά την αφαιρεγκαιότητα. Και τέλος, συμφωνήσαμε ότι η μικρή ομάδα αυτή θα συναντηθεί ε, δύο-τρεις-τέσσερις φορές. Ε, αυτό ήταν ε, καταρχήν ιδέα της κυρίας Μαντουρέλ και της κυρίας Μέρκης. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μία task force. Αυτό μάλλον είναι υπερβολικό βέβαια. Πάντως συμφωνήσαμε να ξανασυναντηθούμε κάποιες φορές ώστε να καταγράψουμε ε, ε, κάποια πράγματα που μάθαμε από την Καλιφόρνια και να τα υποβάλουμε αυτά ε, στην Κομισιόν ή στο Κοινοβούλιο. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα θέματα από τα οποία μπορούμε κάτι να μάθουμε. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν είναι μια ομάδα εργασία η στο κοινοβουλιο να δουμε δηλαδη ποια ειναι τα θεματα απο τα οποια μπορουμε κατι να μαθουμε βραχυπροθεσμα λοιπον ειναι μια ομαδα εργασιας η οποια θα συναντηθεί κάποιες φορές, δεν θα είναι μόνιμη όμως. Εάν συμφωνούμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, ε, τότε θα πρέπει να ε, αδράξουμε κάθε ευκαιρία να διατηρήσουμε την επαφή με τους συνομιλητές που είχαμε στην ε, Καλιφόρνια. Έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ τον είχαμε καλέσει εδώ και σε μια ακρόαση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση αυτή και επίσης ενδιαφέρον ήταν ένα βράδυ που περάσαμε με τις νέες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είδαμε τόση καινοτομία, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βράδυ βραδιά. Ωραία. Έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης. Ε, το συζητήσαμε νωρίτερα από ό,τι λέει. Ε, πάντως το ολοκληρώσαμε. Ε, φτάνουμε τώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην συντάκτρια της νομοδότησης Λένα Εκ για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η δουλειά της Επιτροπής μας ε, σήμερα είναι και αυτή αποτελεσματική, διότι είναι λίγοι βουλευτές εδώ σήμερα, είναι όμως οι πιο αφοσιωμένοι ε, παρόντες. Η μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της ε, είναι ένα από τα θέματα στην Στρατηγική Ευρώπη 2020, την οποία έχουμε συζητήσει στις πολιτικές ομάδες και που έχει συζητηθεί και ε, στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν κάποιες εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 και ε, η Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους είναι μία από τις πρωτοβουλίες αυτές. Ο λόγος που έχουμε την πρωτοβουλία αυτή είναι η εξαιρετική της σημασία για την δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη. Από πολλές απόψεις, αν κοιτάξουμε καταρχήν το θέμα των πρώτων υλών. Ε, θα δούμε πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό. Ε, το 95% ε, του σιδήρου στην Ευρώπη βρίσκεται στο βορρά της Σουηδίας από, ε, τα, από τις σπάνιες γέες Βλέπουμε ότι και αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις νέες τεχνολογίες, ε, για, για γιατρικά μηχανήματα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ε, ε, ανεμόμιλοι κλπ. Οι 10 πιο, που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εισάγονται στην Ευρώπη και για 7 από ε, αυτές εξαρτώμεθα αποκλειστικά από τις εισαγωγές ενώ για τις υπόλοιπες 3 το ποσοστό εισαγωγής είναι 97-98%. Ε, εάν λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, το, ε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε. Θα ανακυκλώσουμε ε, τα υλικά αυτά από τους υπολο, παλιούς υπολογιστές κτλ. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε πρώτες ύλες. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται για να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά και φιλικοί προς το περιβάλλον, διότι αυτά αυτά ε, τα, τα δύο ακολουθούν το άλλο. Άλλος τομέας όπου πρέπει να σκεφτούμε την αποτελεσματικότητα των πόρων είναι η παραγωγή τροφίμων. Για παράδειγμα, ο φόσφορος που είναι ένα από ε, τα τρία βασικά συστατικά των λιπασμάτων. Ε, είναι και αυτό ορυκτό, όπως ε, και ο άνθρακας. Αλλά σε 30-35 χρόνια θα έχουμε έλλειψη. Και εάν δεν έχουμε αρκετό φόσφορο ε, στο χώμα, ε, τα φυτά θα είναι καχεκτικά και κίτρινα και μετά από κάποια χρόνια θα είναι αδύνατον να ε, καλλιεργήσουμε τα εδάφια αυτά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Τι κάνουμε με το φόσφορο σήμερα. Πολλά κράτη-μέρη δεν το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Ε, αυτό τελικά μετατρέπεται σε, ο φόσφορος τελικά μετατρέπεται σε οξύ και αυξάνει την, ε, τα φύκια στη, στα ύδατά μας. Το Λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια γεωργική πολιτική που να είναι αποτελεσματική ω προ ε, την χρήση του φωσφόρου, ώστε να έχουμε φωσφόρο για τουλάχιστον 10 χρόνια παραπάνω. Και αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε με έρευνε ώστε να μπορούμε να βρούμε εναλλακτικού τρόπους ε, παραγωγής ε, τροφίμων ή και παραγωγής λιπασμάτων. Το θέμα αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ε, περιβαλλοντικό, η αποτελεσματικότητα των πόρων είναι και σε μεγάλο βαθμό θέμα ανταγωνιστικότητας ε, και οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά τους πόρους μας από ό,τι κάνουμε σήμερα. Και τώρα με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ε, προγράμματος πλαισίου 7 και που θα ε, αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα έγγραφα για το πρόγραμμα πλαίσιο 8 ε, θα πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και με την ε, Ευρώπη 2020 ε, με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες και να τα συνδυάσουμε αυτά και με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα προβλήματα, θα πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία, ε, θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα στους τομείς αυτούς και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ε, τι εργαλεία έχουμε για την καινοτομία. Υποθέτω ότι όλοι θα χρειαστούμε τρόφιμα στο μέλλον, όπως και ε, αυτοκίνητα, μπαταρίες, για όλων των ειδών τα μηχανήματα και θα χρειαστούμε και ιατρικά μηχανήματα στα νοσοκομεία. Όπως είπα, υπό το φως της ε, ε, δημογραφικής εξέλιξης στον κόσμο, με άλλα λόγια την αύξηση του πληθυσμού, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί ως προς τους πορούς από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Τα προβλήματα όμως τώρα γίνονται πολύ πιο επιτακτικά. Αυτά λοιπόν ε, είναι λίγο πολύ τα θέματα που θα περιέχει η γνωμοδότησή μου. Επίσης, ακούω ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση ή πρόταση της Κομισιόν τον Αύγουστο. Ίσως λοιπόν να είναι χρήσιμο να συνδυάσουμε τις εργασίες που θα έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στην συνεδρία των συντονιστών, κύριε Πρόεδρε. Το τι θα κάνουμε τελικά. Πάντως, ε, περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. συνάδελφος Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσον αφορά το έγγραφο της Κομισιόν. Ε, σημείωσα το περιεχόμενο, ωστόσο, δυσκολεύομαι να καταλάβω ε, τι ακριβώ προσπαθεί να κάνει εδώ η Κομισιόν. Οι πόροι είναι μια πολύ γενική έννοια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο ακριβή ορισμό. Υπάρχουν γεωργικοί πόροι, υδάτινοι πόροι, πόροι στην αλία κλπ. Νομίζω ότι είναι πολύ ευρία η έννοια αυτή. Όσον αφορά τους ορυκτούς πόρους, Ε, αναρωτιέμαι λίγο, διότι έχουμε ήδη το σχέδιο του κυρίου Μπιουτικόφερ. Ε, και δεν βλέπω το λόγο να ε, έχουμε δύο διαφορετικές εκθέσεις για το ίδιο θέμα. Επίσης, όσον αφορά τους γεωργικούς πόρους ε, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Για παράδειγμα, τα Ολικά πάρκα στη Γερμανία με κάνουν να αναρωτιέμαι, διότι βλέπουμε χρήση των πόρων, ε, κατά τη γνώμη μου όμως όχι αρκετά αποτελεσματική. Επίσης ε, σημαντικό είναι για μένα να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά ε, τους γεωργικούς πόρους και τους υδάτινους. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. Στην Πολωνία με το νερό και στο σύνολο της Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος ότι θα δούμε δραματικά γεγονότα στην Παλαιστίνη. Υπάρχει λειψιδρία και στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας. Τι θα συμβεί λοιπόν. Αν ε, ε, κατασκευαστεί ένα ε, φράγμα στον ήλιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολέμους ε, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι το ένα θέμα που ήθελα να αναφέρω. Το άλλο είναι το εξής. Πώ μετράμε του πόρους. Δεν υπάρχουν εδώ σχετικές προτάσεις τη Κομισιόν. Είναι πολύ γενική η πρόταση, είναι πολύ γενικές οι έννοιες που χρησιμοποιούνται. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους μας, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας. Κατά τη γνώμη μου, ακριβώς αυτές οι προτεραιότητες είναι σημαντικές ε, και αυτό λείπει από το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον ε, διάβασα το, την πρόταση της Κομισιόν. Σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες ε, που αφορούν την πρόταση αυτή. Και εγώ θα ήθελα να σας προειδοποιήσω, βλέπουμε εδώ υπερβολική αισιοδοξία. Σημαντικό είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους αλλά και το τι θα κάνουμε με τα απόβλητα κατά τη διαχείριση των πόρων. Ε, σημαντικό είναι η χρήση των πόρων ε, να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχουμε ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων ε, στο φυσικό περιβάλλον στις διάφορες χώρες και ε, τι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Ε, να μην ξεχνάμε ότι η υψηλή τιμή των πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό των κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων από τη χρήση αυτών. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την ε, πλήρωση των στόχων ε, για τις εκπομπές μέχρι το 2050. Σημαντικό είναι να γίνει αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, και αυτών που προέρχονται από την Κίνα και την Κορέα. Τελικά θα πρέπει να αλλάξουμε τη στάση των καταναλωτών, ε, τους τρόπους παραγωγής, ε, αλλά να εξετάσουμε και τη χρήση των δημοσίων πόρων. Όσον αφορά νέους πόρους, όπως είναι το αέριο αποσχιστόλιστο, θα πρέπει και αυτούς τους πόρους να τους εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό νέες τεχνολογίες. Όπως είναι η... η αποθήκευση, η δέσμευση του, του άνθρακα. Ε, υπάρχουν πάντα αισιόδοξα και απεσιόδοξα σενάρια. Θα πρέπει να τα λάβουμε όλα μας υπόψη. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εξέλιξη των τιμών για την ενέργεια και για άλλους πόρους. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της Κομισιόν. Ελπίζω ότι τα θέματα που θα θυχτούν ε, στην έκθεση θα μας βοηθήσουν να ε, εκμεταλλευτούμε πιο ε, αποτελεσματικά τους πόρους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπίτικοφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τη βασική προσέγγιση στο θέμα αυτό, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Εκ. Πολύ σύντομα λοιπόν για κάποια σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι έχουμε εδώ μια καλή ευκαιρία να προωθήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του του τρόπου παραγωγής μας. Ε, η γενική κατανόηση δηλαδή ότι θέλουμε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, ότι χρειαζόμαστε τρόπους παραγωγής αποτελεσματικούς ως προς τους σπόρους, Ε, αυτή συμπεριλαμβάνει ότι ακόμα και ε, οι ύλες που σήμερα θεωρούνται απόβλητα θα πρέπει να αναγνωριστούν ως πόροι. Δεύτερον, Πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ιδιαίτερο καθήκον. Ε, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να εισάγει τόσες πρώτες ύλε όσο εμείς, ε, αν το υπολογίσουμε αυτό ε, ανακεφαλή ε, κάθε χρόνο. Η Ευρώπη λοιπόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πρώτων υλών και γι' αυτό η ευρωπαϊκή οικονομία ε, μπορεί να υποφεληθεί ιδιαίτερα από αποτελεσματική χρήση των πόρων αυτών. Τρίτον, σημαντικό είναι να έχουμε αξιόπιστες μεθόδους κατά τον υπολογισμό των πόρων. Αυτό υπόθηκε ήδη. Και πιστεύω ότι χωρίς ε, σωστούς ε, υπολογισμούς ε, μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να πετύχουμε τους πόρους ακόμα και αν έχουμε καλές ρυθμίσεις. Θα θεωρούσα καλό στην ε, έκθεση αυτή να αναφέρονται οι πόροι που δεν τονίζονται τόσο πολύ στη δική μου έκθεση, συμφωνώ δηλαδή με αυτό που υπόθηκε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε σαφώς μέσα τα οποία θα είναι χρήσιμα και να λάβουμε υπόψη μας και την πτυχή στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την κοινωνική διάσταση. Πιστεύω ότι δεν θα προοδεύσουμε αποτελεσματικά εάν η αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, αντίκειται τελικά στην, ε, στη, στους κοινωνικούς μας ε, στόχους. Και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της τυποποίησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των πόρων. Ε, είναι ένα... Ε, εδώ βλέπουμε ότι ε, διασταυρώνονται δύο θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ, Κομισιόν. Α, ζητάει κάποιος ακόμα το λόγο. Παρακαλώ. Κομισιόν, παρακαλώ. Ο κύριος Ντάνιαν. Τζόνσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ο κύριος Τζόνστον. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω σήμερα και να παρέμβω όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Βασικά, νομίζω θα πρέπει αυτό να το δούμε ως την αρχή μιας διαδικασίας της πρωτοβουλίας Ναυαρχίδας που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο φέτος, διότι περιγράφει το πρόβλημα, ε, περιγράφει το ποιοι πόροι καλύπτονται, ε, πρόκειται για φυσικούς πόρους, κάθε είδους πόρους μάλιστα, και προσπαθεί να θεσπίσει μια διαδικασία που εξετάζει το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη πολιτικό πλαίσιο. Έχουν εξεταστεί διάφορες πρωτοβουλίες, δύο έχουν υιοθετηθεί ήδη με μακροπρόθεσμους στόχους και δύο άλλες σημαντικές που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Έχουμε το, την Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές και αργότερα φέτος θα έχουμε τις, μακροπρόθ, τις, τις, μακρο, τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για την ενέργεια και έναν οδικό χάρτη προς την ευρωπαϊκή οικονομία που είναι αυτάρκης στους πόρους. Βασικά λοιπόν είναι η αρχή της διαδικασίας σηματοδοτεί το πλαίσιο και τους στόχους, αλλά αφήνει τις λεπτομέρειες να συμπληρωθούν από πρωτοβουλίες που θα έρθουν αργότερα. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην επάρκεια των πόρων, ε, ένα, μια μελέτη που θα ε, έρθει αργότερα φέτος. Ορισμένα μέλη ήδη το ανέφεραν τη μέτρηση. Πώς μετράμε δηλαδή την, απο... την επάρκεια των πόρων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον θα αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αυγούστου, γιατί διαφορετικά θα μπορούμε να κρίνουμε την πρόοδό μας, να δούμε δηλαδή πώς βελτιώνουμε τη χρήση των πόρων εντός της Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για σήμερα. Α, η κυρία Εκ και πάλι παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω και ευχαριστώ μάλλον όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Έχουμε κάποιες κοινέ ανησυχίες και μία κοινή γραμμή για αυτό το κείμενο. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπα νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, ότι πιστεύω πως οι συντονιστές θα πρέπει να σκεφτούν το γεγονός ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης σε λίγες εβδομάδες για το ίδιο θέμα, για να μην γίνει η επικάλυψη της εργασίας. Θα πρέπει αυτό να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα το χειριστούμε σε επίπεδο συντονιστών. Ευχαριστώ. Ωραία. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν να έχουμε μια ιδέα σχετικά με το τι θα κάνουμε, όχι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά να έχουμε μια ιδέα σχετικά με το ποια θα είναι η σχετική λύση. Ε, ωραία. Ε, αν συμφωνείτε θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα λοιπόν. Ατζέντα για νέε δεξιότητε και θέσει εργασία. Η Νίκη Τζαβέλα είναι τάξη τη νομοδότηση. Έχει τον λόγο, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, first of all, I would like to Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και... Ε, ε, καταρχήν, συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάστος για την εξαιρετική της έκθεση που καλύπτει εκτεταμένα την νέα... τη νέα ανακοίνωση περί δεξιοτήτων και θέσεων απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. οι πατρίες που έχω να κάνω ως εισηγήτρια και ως ε, μέλος της Επιτροπής Ήτρε είναι οι εξή. Καταρχήν, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στις πολιτικές διαβίου κατάρτισης ώστε να λειτουργήσει καλύτερη αγορά εργασίας μας. Πρέπει να τονίσουμε την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων ε, της, ε, στην πληροφορική. Δεύτερη παρατήρηση πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων μέσα, ανάμεσα στα κρατη Γι' αυτό και θα πρέπει να ενεργήσουμε προς τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας που θα είναι υπεύθυνη για την ε, διοχέτευση εργατικού δυναμικού προς τις χώρες που το χρειάζονται υποστηρίζοντας έτσι με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία την αγορά εργασίας. Επίσης πρέπει να εγγυηθούμε ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Στην ανακοίνωση υπάρχει μια προτινόμενη μείωση του εργατικού κόστους που θα κινητοποιήσει και θα οθήσει την ανάπτυξη. Ωστόσο, η μεγάλη φορολογία στην ενέργεια ή στις ε, ε, εκπομπές για να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων για τις κοινωνικές περιοχές θα αφήσουν τις επιχειρήσεις με άνισο βάρος και επίσης θα οδηγήσουν σε ψηλό κόστος ε, παραγωγής και έτσι θα καταστρέψουν θέσεις παρά θα ε, ε, έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ήδη τονίζεται η δυνατότητα αυτή στην γνωμοδότηση και γι' αυτό τονίζω στη δική μου γνωμοδότηση ότι η απώλεια από τις κοινωνικές παροχές θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από μεθόδους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χαμηλότερο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ. <clears throat> Gracias, señor Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε για μια έκθεση πολύ ε, κέρια για το μέλλον της Ευρώπης, για το μέλλον των νέων μας, που είναι αυτό της υπήρου μας. Κατά τη γνώμη μου, το να βελτιωθεί η προετοιμασία και η δεξιότητα όλων των εργαζομένων είναι η μόνη λύση προς μια μεγαλύτερη απασχόληση και καλύτερης ποιότητας. Η καλύτερη κατάρτιση είναι ένα βασικό βήμα για να βγει η Ευρώπη από την κατάσταση αυτή της κρίσης στην οποία βρίσκεται, για να μπορέσει να εγγυηθεί την ανάπτυξη των επόμενων δεκαετιών. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρώπη να βασιστεί σε μια Ευρώπη που βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία. Και αυτό και σε στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020, ακριβώς για να αντιμετωπίσει την ε, νεανική ανεργία θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε προγράμματα κατάρτισης, ενημέρωσης ε, για να μπορέσουμε έτσι τα κριτήρια αυτά να είναι κριτήρια στη βάση της πολιτικής απασχόλησης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα η ομάδα των σοσιαλιστών θα δώσει την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην ανάπτυξη της ατζέντα για τις νέες δεξιότητες ε, έτσι ώστε τα προγράμματα να χρηματοδοτούνται καταλήλως. Είναι αναγκαίο λοιπόν να συνεχίσουμε στο μέλλον. Όπως είπε ακριβώς και η προλαλή σας, πρέπει πραγματικά να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να μπορούμε και να δημιουργήσουμε απασχόληση, ιδιαίτερα για τα εκατομμύρια νέων που βρίσκονται στην ανεργία. Ευχαριστώ. Η κυρία, Η ε, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για το κείμενο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει να πω ότι διστάζω πάρα πολύ για το σημείο 3. Θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει μήπως μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οργάνωση για ελεύθερες θέσεις απασχόλησης. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι αρμοδιότητα η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε ιδιωτικούς φορείς, ή ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να φροντίσουν οι δημόσιοι οργανισμοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα να έχουν ένα τμήμα για θέσεις απασχόλησης σε διεθνές επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια σήμερα. Έχουν την τάση να δουλεύουν με την πολυτοπική αγορά, με τις θέσεις απασχόλησης τοπικά μόνο και να μην κοιτάνε τι υπάρχει στην Ευρώπη ολόκληρη. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο 3 θα ήθελα να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να γίνεται αυτή η δουλειά, να αναλάβει κάποιος αυτό το καθήκον. Και δεν ξέρω μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία για αυτό το σκοπό. Δεν ξέρω. Τώρα για το σημείο 5. Γίνεται συζήτηση για μείωση του κόστους εργασίας. Μιλάμε για τα, την απώλεια εσόδων, για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Και εδώ πάλι τα κράτη-μέλη πρέπει να λειτουργούν καλά. Συμφωνώ απόλυτα για το ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και ότι πρέπει, ναι, συμφωνώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα ήθελα να υπάρχει και κάτι άλλο που να μιλάει για την καινοτομία και για το τι κάνουμε μετά. Εκεί δηλαδή που είμαστε αδύναμοι. Έχουμε συχνά πολύ καλά προϊόντα, τα οποία αγοράζονται στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Νότια Κορέα, Βραζιλία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, που θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν κατασκευαστεί εδώ στην Ευρώπη. Είναι κρίμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μπει κάτι εδώ υπέρ τη καινοτομία σε εμά και το τι κάνουμε με αυτήν στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπρεζίνα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι ικανοποιημένος που ασχολείται με αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν είμαι ικανοποιημένος για αυτό που έθιξε η κυρία Εκ, ότι δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος οργανισμού. Η προλαλήσεσαι... Ε, έκανε διάφορες παρατηρήσεις και συμφωνώ για το ότι είναι ένα θέμα ευθύνης των μεμονωμένων κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι καθένας από εμά έχει ένα τμήμα της ευθύνης για την ε, απασχολησιμότητά του. Εάν σήμερα το προφίλ της ε, απασχόλησης για πολλούς ε, άνεργους είναι τέτοιο που για τις ε, περισσότερες φορές ας πούμε, μπορούν να απασχοληθούν στην ε, κρατική διοίκηση και μιλώ για τομείς που είναι εκτός της αγοράς εργασίας, εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε για ευθύνη καθενός από εμά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν στον τομέα της ε, κατάρτισης ε, των φοιτητών αλλά και των γονέων για την επιλογή. για να μπορούν δηλαδή να, να καταρτιστούν για θέσεις που ζητά η αγορά εργασία. Ο συνάδελφο Όντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να προτείνω να σκεφτούμε μια καλύτερη συμμετοχή, μάλλον εμπλοκή του κοινωνικού διαλόγου στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Βέβαια, κάθε κράτο μέλο έχει το δικό, και στι οργανώσει κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στα, στους και του εργοδότε, αλλά νομίζω πω είχε ώρα η Κομισιόν να μπορέσει να απευθύνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνη στο κοινωνικό διάλογο σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλα τα θέματα, πολιτικές κατάρτισης, ε, Ποιο ε, μπορεί να ξέρει καλύτερα τι είναι καλό για τη χημική βιομηχανία, α πούμε, από τους χημικούς μηχανικούς, το ίδιο για την αυτοκινητοβιομηχανία, για τις ασφαλίσεις, για τις τράπεζε, Έχουμε μέσα στην συνθήκη που να επιτρέπουν σε ευρωπαϊκή κλίμακα να έχουμε ένα κοινωνικό διάλογο και να έχουμε και συλλογικές ε, συμβάσεις που είναι η αρχή της, ε, του σχηματισμού ενός ε, κοινωνικού δικαίου εργασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα την ευελιξασφάλεια για την οποία χαίρομαι που η Κομισιόν το ξαναβάζει αυτό προς μελέτη και να μπορέσουμε να φτιάξουμε έτσι ένα σημαντικό διάλογο σε επίπεδο ευρωπαϊκό που υπάρχει, αλλά που θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο. Ο συνάδελφος Πίτικοφερ. Κόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης και να κάνω κάποιες προσθήκες στο σημείο 2 Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό να αναφερθούμε στα ICT, στις ε, τεχνολογίες ε, ε, πληροφορικής και επικοινωνίας και πιο κάτω θα ήθελα να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις δύο συναδέρφων. Δεν είμαι βέβαιος ότι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Στο σημείο 4 βρίσκω σημαντικό να αναφερόμαστε στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και να αναφέρουμε ρητά τις δεξιότητες. Ιδιαίτερα έχοντας κατά νου το ερώτημα ποιο, τι ρόλο θα παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια κατά την πρόθεση της καινοτομίας. Να μην επιτρέψουμε, να το πω έτσι, να μιλούν όλοι για μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά στα σημεία όπου πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διασφάλιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, κατά ε, την έρευνα κτλ, να μην ε, μπορούμε να προσελκύσουμε την προσοχή του κόσμου. Και επίσης στο σημείο 5 θα ήθελα να προσθέσω να μην αναφέρουμε αποκλειστικά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας ε, ως μέτρο, αλλά και την κοινωνική προστασία των ε, εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για, την, ε, για το σχέδιο Ε, της ε, γνωμοδότησης. Με χαρά σημειώνω ότι αναφέρεται ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για να τονίσουμε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τομέα και όσον αφορά την ε, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ε, εργαζομένων. Η ε, εργαζόμενοι πρέπει να έχουν όχι μόνο γνώσεις, θα πρέπει να έχουν και δεξιότητες. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, ε, τέτοιες επιχειρήσεις, ε, γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η διαβίου μάθηση για τους εργαζομένους αυτούς. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εκπαίδευση που προτείνεται εδώ είναι πολύ σημαντική. Θυμάμαι μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας, ε, κατά την οποία υπόθηκε ότι η Ευρώπη χάνει σε σχέση με τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες, διότι εκπαιδεύουμε επιστήμονες, ε, όχι όμως επιχειρηματίες. Αυτή είναι η διαφορά με τις Ηνωμένε Πολιτείε και νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδέα από τις Ηνωμένε Πολιτείε και να ε, να βοηθούμε στην ε, δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και ε, γίνονται τελικά επιτυχημένοι οικονομικοί παράγοντες. Η εκπαίδευση των εργαζομένων δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές γνώσεις. Θα πρέπει να στοχεύει και σε μια πιο αθερετική σκέψη. Η δημιουργικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα ε, και γι' αυτό θεωρούνται οι δημιουργικοί ε, ε, εργαζόμενοι ιδιαίτερα πολύτιμοι. Χρειάζεται η Ευρώπη περισσότερους ε, εργαζομένους ε, στους τεχνικούς τομείς, ε, χρειάζεται όμως και περισσότερες επιχειρήσεις στην Πολωνία, στην πατρίδα μου. Εκπαιδεύσαμε ανθρώπους που όμως ε, είχαν πιο πολύ ακαδημαϊκές και, τεχνικές, ε, και θεωρητικές γνώσεις παρά τεχνικές στην πράξη. Και ε, έτσι έχουμε αμελήσει την εκπαίδευση των, έχουμε παραμελήσει των ανθρώπων στους τεχνικούς τομείς. Θα πρέπει αυτό το έλλειμμα να το καλύψουμε. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τη διάγνωση του Πιέρο Είπε ότι ο κοινωνικός ε, διάλογος είναι πολύ σημαντικός, είναι απαραίτητος κατά τη γνώμη μου. Αυτό πράγματι ισχύει. Και είναι σημαντικό Ε, να ζητήσουμε και την γνωμοδότηση, για παράδειγμα, των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ε, Πολωνία. Είπατε ότι η γνωμοδότηση της Κομισιόν είναι καλή. Το σημαντικό όμως είναι πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη οι ιδέες αυτές. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο κοινωνικός διάλογος με τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι κανείς εδώ από την Κομισιόν? Θέλει να πάρει κανείς το λόγο από την Κομισιόν, παρακαλώ. Yeah, thank you Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε πολύ για την γνωμοδότησή σας που στηρίζει την Κομισιόν προκειμένου Επίσης σας ευχαριστούμε και για την στήριξή σας όσον αφορά το προσωπικό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση. 23 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα είναι άνεργοι. Η μυρίσια διάταξη θέτει διάφορες προτεραιότητες για τη βελτίωση της αγοράς απασχόλησης με την ευελιξία και την ασφάλεια, με τις δεξιότητες, με την βελτίωση των συνδικών εργασίας και κυρίως με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, όπως είπα πριν, 23 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στην ανεργία και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα Ορισμένου τομεί. Από την άλλη μεριά, για ορισμένες δεξιότητες δυσκολευόμαστε να βρούμε προσωπικό. Οπότε η ανάπτυξη δεξιοτήτων και το τέριασμα των αναγκών με την προσφορά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Να αναπτύξουμε δηλαδή τις σωστές δεξιότητες, αυτές που χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω και το εξή η εφαρμογή της πρωτοβουλίας έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπως λέτε κι εσείς. Οπότε, το πρώτο τριμερές φόρουμ οργανώθηκε το Μάρτιο που μας πέρασε. Ήδη με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη-μέλη, προκειμένου να έχουμε την συμμετοχή όλων στις πρωτοβουλίες για τις πολιτικές ευελιξίας και ασφάλειας για την εργασία. 13 Νοεμβρίου έχουμε και μια διάσκεψη πάλι για το ίδιο θέμα με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν το ποια στιγμή έρχεται η έκθεση αυτή στο προσκήνιο, καταλαβαίνετε ότι θα συνεισφέρει πάρα πολύ και στην διάσκεψη αυτή του Νοεμβρίου. Περιμένουμε την τελική εκδοχή της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Τζαβέλα τώρα έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το σημείο αριθμός 1. Συμφωνώ με τις προτάσεις και τις συστάσεις που έκαναν οι συνάδελφοι όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρόεδρε, διαπιστώνω όμως ότι οι περισσότεροι από εμά επικεντρωνόμαστε στο σημείο 3, εκεί δηλαδή που εγώ προτείνω την πανευρωπαϊκή υπηρεσία. Είχαμε το ελεύθερο κίνημα μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία. Μεγάλο εμπόδιο. Όπως και να έχει όμως το πράγμα. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης προσπαθεί να διευκολύνει την κινητικότητα. Συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι σε πολλές χώρες μέλη θέλουν διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένες ε, δεξιότητες. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει υπογράψει με την Πολωνία διμερή συμφωνία πάνω σε αυτό και η Αυστρία. Αυτό δηλαδή που εγώ ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή είναι ότι το βλέπω να έρχεται. Αν θέλουμε μία ενιαία αγορά, θα έχουμε και μία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μία ενωμένη ενιαία. Τώρα, αν δεν υπάρχει ένας κεντρικός ευρωπαϊκός οργανισμός που το κάνει, εντάξει, ας δούμε τι άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ιδιωτικέ υπηρεσίες. Αλλά έτσι και αλλιώς η κεντρική διεύθυνση θα πρέπει να έρχεται από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ και τον κύριο Πατικόφερ πάντα όταν κάνει σχόλια για την κοινωνική προστασία. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι διαπίστωσα σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Άντος πριν από ένα μήνα δεν απατώμε, όπου είπε ότι ενθαρρύνει, έτσι είπε, encourage, ενθαρρύνει λοιπόν την κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών μελών. Είτε πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη από κάποιες δεξιότητες εργατικού δυναμικού ή αντίθετα κάποιες άλλες έχουν πλεόνασμα δεξιοτήτων. Αυτό ήταν ένα άλλο σχόλιο που έχω να κάνω όσον αφορά την παράγραφο 3 της εκθεσής μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείνουμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Α, ο κύριος Σόντι, παρακαλώ. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, Πρόεδρε, αλλά ακούγοντας τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω αυτή η μετάφραση, πάντως κατάλαβα ότι είπατε 14 Νοεμβρίου θα είναι η διάσκεψη αυτή και ότι θα είναι μαζί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλή πρόταση, αλλά 14 Νοεμβρίου εμείς έχουμε σύνοδο στο Στρασβούργο. Δεν ξέρω αν σωστά έφτασε η ημερομηνία στα αυτιά μου ή όχι. Ερώτηση προς την Κομισιόν, είναι σωστή η ημερομηνία αυτή? Ναι, ναι, ναι αυτή είναι η ημερομηνία, πράγματι. Είναι Δευτέρα. Äh, Αυτό συχνά είναι πρόβλημα. Το έχω διαπιστώσει επανειλημμένα ότι η Κομισιόν ε, κανονίζει πράγματα όταν ε, βρισκόμαστε εμείς ε, στο Στρασβούρο. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Ο κύριος Σοντή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λέει ότι περιμένει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον προηγουμένως δεν έχει ελέγξει την ημερομηνία. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσε η Επιτροπή να ζητήσει από την Κομισιόν ε, να επανεξετάσει την ημερομηνία για να επιτρέψει τη συμμετοχή ε, στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί, απαντάει ο Πρόεδρος, το θέλει επίσης. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε τότε λοιπόν. Μια επιστολή προς την ε, Κομισιόν. Εγώ ευχαρίστω ε, στέλνω επιστολές. Ε, θέλετε να την ε, διαβάσετε και πριν τη στείλω. Α, βλέπω ότι δεν χρειάζεται να την ελέγξετε. Ε, εντάξει. Okay. Damit machen wir das. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Ε, σας παρακαλώ όμως να μεταφέρετε το αίτημά μας αυτό ούτως ή άλλως. η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών 21 Ιουνίου 12 η ώρα. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ε, το αποφασίζουμε λοιπόν. Ε, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι οι πρώτες ύλε. Ε, ο συνάδελφος Μπίτικοφερ είναι αρμόδιος, θα πάρει λοιπόν και πρώτος τον λόγο με μικρόφωνο, Απολύτω επισήμως θα μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν σαφές ότι η προσπάθεια του συναδέρφου Λάγκε να μου αποσπάσει την προσοχή δεν θα ε, πετύχαινε, αλλά σας ευχαριστώ παρόλα αυτά ε, για την ε, καλή σας πρόθεση. Είχαμε μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Κατά την συνάντηση αυτή είχα 30 προτάσεις Ε, για ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Κατά τη δική μου γνώμη ήταν ε, εξαιρετικά επιτυχημένη η συνάντηση αυτή. Δεν υπήρχε πουθενά η εντύπωση ότι υπάρχουν δυσκολίες που δεν μπορούν να λυθούν. Ήταν πολύ επικοδομητικό το πνεύμα. Δεν ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Δεν προλάβαμε να εξετάσουμε όλες ε, τις τροπολογίες. Θα έχουμε λοιπόν ένα δεύτερο γύρο, κατά τον οποίο θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη μου τις ε, παρατηρήσεις τις ε, προτάσεις ε, για προσθήκες ε, κλπ. που ακούσαμε κατά τις συζητήσεις αυτές. Ελπίζω λοιπόν ότι τελικά θα έχουμε μια καλή βάση για την ψηφοφορία. Ε, όσον αφορά τη διαδικασία, έχουμε μία δυσκολία την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήδη έχει ψηφίσει τις τροπολογίες της, ε, έτσι θα ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη ε, κατά την εκπόνηση των συμβαστικών τροπολογιών. Ε, μπόρεσαν να ληφθούν υπόψη. Αυτό δεν ισχύει για την Επιτροπή Περιβάλλοντος όμως ε, και την Επιτροπή Εμπορίου που πολύ λίγο πριν ε, την δική μας ψηφοφορία θα ψηφίσουν τις δικές τους τροπολογίες, νομίζω μία ή δύο μέρες πριν. Δεν μπορώ λοιπόν να εγγυηθώ ότι θα συμπεριληφθούν όλα αυτά στις συμβαστικές τροπολογίες. Και η Επιτροπή ΝΤΕΔΕ έχει υποβάλει προτάσεις. Τελικά μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να ψηφίσουμε μία προς μία τις προτάσεις τους αυτές. Δεν βλέπω όμως να είναι πρόβλημα αυτό, ούτε πιστεύω ότι αυτό είναι άδικο απέναντι στις ε, επιτροπές αυτές που θα γνωμοδοτήσουν. Δεν θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία προς μία τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αρκούν αυτά που σας είπα και περιμένω να ακούσω παρατηρήσεις ή προτάσεις των συναδέρφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει κάποιοι τον λόγο. Πρώτα η σκιώδης ε, η κυρία κυρία Σκογ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο εισηγητής, είχαμε πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά την στρατηγική για, τα, για τις πρώτες ύλες. Είχαμε ήδη την πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών και είδαμε σε μεγάλο βαθμό συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες συμβαστικές ε, τροπολογίες. Η πολύ καλή αυτή έκθεση καλύπτει πολλά σημαντικά θέματα. Όσον αφορά τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες, Είναι πολύ ευρία η στρατηγική αυτή. Έχει να κάνει με τον εφοδιασμό πρώτων υλών προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ασχολείται όμως ε, και με ε, την εξόριξη, ε, με την ανακύκλωση κλπ. Ε, ασχολείται δηλαδή και με τα θέματα και με τις περιβαλλοντικές πτυχές. Επίσης ε, η ε, πολιτική πρώτων υλών πρέπει να τη δούμε και υπό το μάτι της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης, της σχέσης μας δηλαδή με τον γύρο κόσμο. Σήμερα Είχαμε και την έκθεση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, στην ημερήσια διάταξη, η οποία ε, και αυτή η γνωμοδότηση συνδέεται στενά με την έκθεση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Θεωρήσαμε ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν ήταν υπερβολικά στενή Ε, ήταν κάτι που μάλλον είχε εκπονηθεί με βάση τον κατάλογο για, ε, των σπανίων γεών, ε, αλλά εμείς θέλουμε κάτι πιο ευρύ. οι συμβαστικές τροπολογίες λοιπόν περιλαμβάνουν αυτή την ευρεία στρατηγική, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχουν κάποια θέματα, αυτά που έχουν να κάνουν με την αηφορία, αλλά και την ε, δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ε, την δημιουργία ευημερία, την κάλυψη των δικών μας αναγκών ε, όσον αφορά τι τις πρώτες στην Ευρώπη. Υπάρχει βιομηχανία πρώτων, υπάρχει τομέα ε, πρώτων υλών εντός ε, των ε, σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να λύσουμε τα θέματα μεταφοράς, της έρευνας και της ανάπτυξης Θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά ε, πέρα από τα θέματα ε, ε, ανακύκλωσης περιβάλλοντος κλπ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τώρα λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές αυτές στις συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως, όπως υπόθηκε, συνεχίζουμε τις εργασίες μας πάνω στις συμβαστικές τροπολογίες. Όσον αφορά τι διατυπώσει που αφορούν την πολιτική ανάπτυξη, για μα είναι σημαντικό να παραμείνει εδώ το εμπόριο, η διατύπωση ε, για, το εμπόριο. Υπάρχει συμβαστική τροπολογία που πηγαίνει προ την αντίθετη κατεύθυνση ε, ε, κατόπιν αιτήματος σε άλλων πολιτικών ομάδων. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και ότι ο εισηγητή Beauty Κόφερ ε, θα ε, λάβει αρκετή στήριξη για τις, προτάσεις του ακόμα και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ και πάλι τον συνάδελφο Μπουδικόφερ για την δουλειά που έχει κάνει. Γενικά μιλώντας, πιστεύω ότι έχει συμπεριλάβει πολλά θέματα που θέλαμε και υπάρχει συνοχή τώρα στο κείμενό του όσον αφορά τις Πανιζιές. Θέλω να αναφερθώ σε μια συμβαστική τροπολογία μου τώρα, την οποία δεν βλέπω. Ένα μέρος τουλάχιστον της τροπολογίας. Πρόκειται ιδιαίτερα για τα μέταλλα, στο τέλος της συμβαστικής τροπολογίας, ιδιαίτερα τα μέταλλα. Σίγουρα αναφέρονται διάφορες πρώτες ύλες στην αρχή της τροπολογίας, στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι το να γίνεται ειδική μνήμα σε μία από τις πρώτες ύλες τόσο βασική όπως είναι τα μέταλλα, είναι κάτι που χρειάζεται. Παίζουν σημαντικό ρόλο Επίσης, αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ανάλογα με τη χώρα, κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονται σε μία πρώτη ύλη ή σε μια άλλη πρώτη ύλη, είτε ανάλογα με τη ζήτηση, είτε ανάλογα με την προσφορά. Για άλλες χώρες, ας πούμε, το ξύλο είναι πρωταρχική σημασίας, γιατί έχουν, προσφέρουν ή άλλες πρώτες ύλες, τέλος πάντων. Στην συμβαστική αυτή τροπολογία λοιπόν το αναλέμε particularly metals, τροπολογία αριθμός 4. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα γιατί γίνεται διάκριση σε σχέση με άλλες πρώτες ύλες και πλήττονται έτσι τα απόλυτα θεμητά συμφέροντα ορισμένων χωρών που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέταλλα αλλά ίσως για κάποια άλλη προτήλη. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλές οι συμβαστικές τροπολογίες σίγουρα. Οι τροπολογίες έχουν βελτιωθεί πολύ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανακύκλωση. Και όσον αφορά τη χρήση ιδίων πρώτων αναφέρεται και η ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι οι υπάρχουσες διατάξεις ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε κατά των ε, νέων ε, ρυθμίσεων. Πιστεύουμε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία απλά πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα. Μπορεί κατά εξαίρεση να είναι απαραίτητες κάποιες νέες ρυθμίσεις. Ε, αυτό όμως θα πρέπει να ακολουθήσει μια ε, εντελεχή μελέτη επιπτώσεων ε, για τον τομέα στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι αναφέρεται πολύ σωστά ο ρόλος της εξωτερικής πολιτικής διότι αυτή η εξωτερική πτυχή της, ε, των πρώτων υλών είναι πολύ σημαντική. Κυρία Η, κυρία Τσαβέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πουτικόφερ για την ε, εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει στην έκθεση αυτή. Η αύξηση στη ζήτηση πρώτων υλών παγκοσμίω σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει με συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει απειλή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και γι' αυτό και χαίρομαι που βλέπω ότι πρώτα απ' όλα υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει η έρευνα και η καινοτομία προκειμένου να αναπτύξουμε κατάλληλες τεχνολογίες για ε, μεθόδους ε, βιώσιμης παραγωγής. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, Όσον αφορά τώρα την διπλωματία των πρώτων υλών, είναι και αυτή πολύ σημαντική γιατί έτσι διασφαλίζουμε την, προήθεια, την προμήθεια μέσω συνεργασίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ε, ιδιαίτερα απέναντι σε χώρες όπως η Κίνα. Από εκεί και πέρα τώρα. Και θα ήθελα ο κύριος Μπουτικόφερ να μας ε, επιχειρηματολογήσει σχετικά. Γιατί στη συμβιβαστική τροπολογία τις συμβαστικές τροπολογίες λέμε πόσο σημαντικός είναι ο ίδιος έλεγχος όσον αφορά το εμπόριο με αυτές τις χώρες. Γιατί, γιατί πρέπει να έχουμε μια ήπια προσέγγιση απέναντι σε αυτές τις χώρες στην αρχή. Μια που πρόκειται για, μια νέα αρχή σχέσεων με χώρες που παράγουν πρώτες ύλες. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει, βοηθώντας τις χώρες αυτές, ώστε να έχουν μια αϊφόρα ανάπτυξη και αυτό μέσα από ε, συμφωνίες που χαίρουν διαφωνίας και από τις οποίες έχουν να κερδίσουν και δύο πλευρές. Στηρίζω επίσης την πρόταση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητες εξόριξης σε διάφορες τέτοιες χώρες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτών τηρώντας και σεβόμενοι περιβαλλοντικές, εργασιακές και κοινωνικές προδιαγραφές. Και θα ήθελα αυτό να συμπεριλαμβάνεται όντω στην έκθεση αυτή. Και πάλι ευχαριστώ και συγχαρητήρια τον εισηγητή, στον κύριο Μπουτικοφέρ. Miss Hall. Thank you. Um, first of all, κυρία Χολ, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για αυτά που είπε ότι λαμβάνει υπόψη και άλλες επιτροπές. Την Αναπτυξιακή Επιτροπή, για παράδειγμα, όπου και εκεί παρακολουθούμε αυτή την ε, έκθεση. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς, να έχουμε μια συνοχή όσον αφορά την πολιτική μας για τις πρώτες ύλες. Και γι' αυτό χαίρομαι για τις τροπολογίες που βλέπω εδώ μπροστά μου, που ζητούν μια τέτοια συνοχή στην πολιτική μας. Ιδιαίτερα συμφωνώ με τι τροπολογίες εκείνε, οι οποίες υπογραμμίζουν το πόσο μεγάλη σημασία έχει η συνοχή αυτή για την ανάπτυξη. Και τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταχειριζόμαστε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες διαφορετικά από ό,τι τις αναδυόμενες οικονομίες. Αναγνωρίζοντας δηλαδή τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πρώτες ύλε υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης τέτοιων χωρών, ιδιαίτερα εφόσον αυτές έχουν την δυνατότητα να τις επεξεργαστούν και όχι μόνο να τις εξάγουν. Ελπίζω η πτυχή αυτή να ληφθεί υπόψη ως τμήμα της ε, προσέγγισης πολιτικής συνοχής. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Χαίρομαι πολύ επίσης που σε πολλές τροπολογίες υπογραμμίζεται η σημασία που έχει η εκ νέου χρήση και η ανακύκλωση των πρώτων υλών. Γιατί όντως είναι κλιματικό να χάνονται ε, σε χωματερές πρώτες ύλες, τόσο πολύτιμες πρώτες ύλες. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφάνεια. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι οι εταιρείε εξόριξης δημοσιεύουν τα έσοδα τα οποία έχουν αναχώρα ώστε οι διαδικασίες εξόριξης πρώτων υλών να μην γίνονται με τρόπο όπου διάφορα καθεστώτα διαφθαρμένα υποφελούνται από αυτές. Και θα έπρεπε να έχουμε τους ίδιους κανόνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελειώνω ευχαριστώντας για άλλη μια φορά τον εισηγητή για το έργο του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με μερικές καλές συμβαστικές τροπολογίες. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ. Πράγματι, όντως, ε, δεν υπάρχει αρκετό χώρο για να συμπεριληφθούν ε, προτάσει και από άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Είμαι κι εγώ από την ΕΜΒΗ συνεισηγήτρια και μπορώ κι εγώ να πω κάτι λοιπόν από αυτού. Ο κύριος Μπιτικόφερ έχει ετοιμάσει μια καλή έκθεση και τον συγχαίρω γι' αυτόν. Στηρίζουμε όλα όσα ανέφερε και προλαλήσει. Είναι πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για στρατηγική για τις πρώτες ύλε να βλέπουμε το θέμα ευρύτερα και να μην το περιορίζουμε μόνο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαρά βιομηχανική μας πολιτική. Θα υποβάλουμε τροπολογίες και σας το λέω από τώρα. Οι σημερινές βιομηχανικές ε, πρώτες ύλε μπορεί να μην είναι οι ίδιες και στο μέλλον, να μην είναι και στο μέλλον δηλαδή εξίσου σημαντικές, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το έχουμε δει αυτό με τα καύσιμα, για παράδειγμα, ότι έχουν γίνει αλλαγέ. Χρησιμοποιούσαμε κάποιε πρώτε ύλε, τώρα προτιμάμε άλλε. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποια μέταλλα, μετά από μερικά χρόνια να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να χρησιμοποιούμε περισσότερο το ξύλο αργότερα ή να βρούμε άλλα φυτικά υλικά τα οποία να θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί και να μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα οποία τώρα ισχύουν και αυτά τα οποία είναι της μόδας σήμερα για τη βιομηχανία. Θέλω επίσης να προσέξουμε και κάτι άλλο. Να μην κοιτάμε μόνο τον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής αυτής για τις πρώτες ύλες, αλλά και τον δεύτερο πυλώνα, αλλά και τον τρίτο πυλώνα και πάνω απ' όλα να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Αντί να εισάγουμε από μακριά, να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη, τι μπορούμε να βρούμε μέσα στην Ευρώπη από πρώτες ύλες και πόσο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Πώς μπορούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποδοτικοί με τα υλικά αυτά και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία τους με τις εφαρμογές δηλαδή που έχουμε. Προσοχή λοιπόν. Όπως έχει συμβεί και με τα απόβλητα και την ιεραρχία τους, έτσι και εδώ πρέπει να έχουμε κάποια ιεραρχία. Δεν λέω ότι πρέπει να την καθορίσουμε από τώρα μια και έξω, αλλά να προσέξουμε, να δούμε από αυτά τα υλικά πού μπορούν να έχουμε τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και ανάλογα με αυτό να δούμε και τη στρατηγική μας. Θέλω και να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ένα σωρό ανακοινώσεις και στρατηγικές ε, αυτή την εποχή. Τι εμβληματικές προτάσεις ή δεν ξέρω εγώ πώς ονομάζονται. Το θέμα είναι όμως ότι από νομοθεσία, από ρύθμιση δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Γι' αυτό και ρωτάω, μήπως θα ήταν καλή ιδέα στην έκθεση αυτή να βάλουμε και κάποιους στόχους κάποια πράγματα που να θέλουμε να πετύχουμε, κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την απόδοση, για παράδειγμα, ή για μια chain of custody, όπου, όπως και με το ξύλο, δηλαδή κατά πόσο τα αυτά είναι υπεύθυνα κοινωνικά. Να συμπεριλάβουμε και κάτι τέτοιο μέσα σε αυτή την έκθεση και αυτό ζητάω από, την, από τον εισηγητή περισσότερη σημασία στα deliverables, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Γκέρεκ. Σας ευχαριστώ. Όταν δει κανείς κανείς την προϊστορία. Όταν δηλαδή εμφανίστηκαν τα πρώτα ανθρώπινα όντα στην γη, είχαμε στην μαδέρα την πέτρα, και, ε, ε, είχαμε το ξύλο μου και την πέτρα ως πρώτες ύλες. Ε, και μετά με την ανάπτυξη προέκυψε το σίδερο, ο χαλκός και ούτω καθεξής τι θέλω να πω, ότι κάθε πρωτήλη έχει το αντίστοιχο, την αντίστοιχη της ενεργειακή ύλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν κάτι είναι μέσα, μένω μέσα στη γη δεν έχει αξία, δεν έχει κέρδος από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ότι η πρωτήλη αυτή υπάρχει. Όταν όμως πρόκειται να εξορίξουμε αυτή την πρωτήλη, τότε ναι, τότε αποκτά αξία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ταξινομήσουμε τις πρωτεσίλες έχοντας υπόψη μας ε, την ε, ενεργειακή τους αντιστοιχεία. Κατά δεύτερο λόγο, και εδώ συμφωνώ με τη συνάδελφο Μέρκης, θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά τον ανεφοδιασμό σε πρώτες ύλες, αυτός ο ανεφοδιασμός αναφέρεται σε ποιες πρώτες ύλες, σε ποιες θα είναι οι απαραίτητες πρώτες με βάση αυτά που χρειάζονται οι κατασκευαστές για την αγορά. Υπάρχει επίσης η καινοτόμα χρήση υλικού στην, ε, από τους μηχανικούς για παράδειγμα. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι πρότυπο, το πρότυπο κατανάλωσης. Διότι το σημερινό μας πρότυπο κατανάλωσης το δεν είναι... Ε, ε, δεν αρκεί όσον αφορά τους πόρους, την ενέργεια, ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να χαράζουμε μία ενεργειακή πολιτική και πολιτική πρώτων υλών, γιατί διαφορετικά στο μέλλον δεν θα έχουμε πόρους για όλη την ανθρωπότητα. Και τέλος, θα ήθελα επίσης να θυμίσω αυτό που υπόθηκε από τον εισηγητή, ότι δηλαδή το θέμα της φορολογίας που συζητείται πολύ για τα περιβαλλοντικά θέματα. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους φόρους επί των εισοδημάτων με τους ενεργειακούς φόρους, γιατί τέτοιου είδους φορολόγηση θα έχει τελικά αρνητικά αποτελέσματα, αρνητικές επιπτώσεις. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αναλύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον συνάδελφο κύριο Μπιτικόφερ θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά του καθώς επίσης και για το γεγονός ότι τις περισσότερες τροπολογίες που υπέβαλα σχετικά με τις σπάνιες γέες τις περιέλαβε στις συμβιβαστικές. Βρίσκω την ευκαιρία να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που βρίσκω ότι σε αυτό το στάδιο της συζήτησης έχουν τη σημασία τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε πού βρίσκεται η Ευρώπη σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού με σπάνιες γέες από την Κίνα. Γιατί το λέω, γιατί πρόσφατα η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι για το δεύτερο μισό του 2011 στις ποσοστώσεις εξαγωγών θα συμπεριληφθούν και τα κράματα τα οποία περιέχουν τουλάχιστον ποσοστό 10% στις σπάνιες γέες. Άρα και γνωρίζουμε ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις των ελήψεων... σε ποιες βιομηχανίες, σε τι ακριβώς γίνεται με την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και της άμυνας. Το δεύτερο είναι ότι επίγει να εξετάσουμε τη δυνατότητα βιώσιμης εκμετάλλευσης εναλλακτικών πόρων σπανίων υγειών εκτός της Κίνας, παράδειγμα την Γρυλανδία, αλλά και να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με τον εντοπισμό εγχωρίων κοιτασμάτων και την ανάπτυξη εγχώριας εξόρυξης, εξευγενισμού και παραγωγής σπανίων γεών, γιατί δεν θέλουμε να διαιωνίσουμε την εξάρτησή μας από τρίτους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η έρευνα και η καινοτομία, η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και η διασφάλιση επαρκούς και υψηλά ειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου βρίσκω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να καταρτήσει μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τις πρώτες ύλε έως το 2050, στον οποίο θα εντοπίζονται πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, απειλές και δυνατότητες στους τομείς των πρώτων υλών και των κρισίμων πρώτων υλών, και με τον οποίο θα βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά ιδρύματα, ώστε να ασχοληθούν με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις επενδύσεις. Ακόμη θεωρώ ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μηχανισμού αποθεματοποίησης, peeling, πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας και ιδίως σπανίων υγεών, ο οποίος θα εγγυάται την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιριών σε στρατηγικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην πράσινη βιομηχανία, τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, τη βιομηχανία άμυνας και τη βιομηχανία υγείας, καθώς και την προστασία από μονοπωλιακές προπιέσεις και αυξήσεις των τιμών. Αυτό με κάποιες προϋποθέσεις φυσικά και ενδεχομένως μέσω συνεργασίας με διεθνείς εταίρους. Να σημειώσω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινες τεχνολογίες όταν οι πρώτες ύλες και ιδίως οι σπάνιες γέες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός υβριδικού αυτοκινήτου ή μιας αναμογεννήτριας έχουν παραχθεί με περιβαντολογικά μη βιώσιμες μεθόδους στην Κίνα. Το περιβαντολογικό αποτύπωμα των πρώτων υλών αλλά και των τελικών τους προϊόντων οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Στη ΣΥΠΑ υπολογίζουν ότι ακόμη και αν ανοίξουν όλα τα ορυχεία σπανίων γεών, θα έχουν ανάγκη από 80 διδακτορικά σε σπάνιες γέες κάθε χρόνο για τέσσερα χρόνια προκειμένου να ανακτήσουν μια ελάχιστη τεχνογνωσία, τεχνογνωσία αξιοποίηση των σπανίων γεών. Στην Ευρώπη έχουμε υπολογίσει τι χρειαζόμαστε. Διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Πώ θα το αναπτύξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Χθε η Επιτροπή οργάνωσε μια σημαντική διάσκεψη για τι σπάνιες Αναρωτιέμαι, είχε προσκληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχαν διάφορε διάφορες προσωπικότητες και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπής πήγε επίτροπη, ε, πρόεδρος των 20 που είναι Ευρωπαίος, όλοι εκφράστηκαν σχετικά με τις πρώτες ύλες, για τις πρώτες Πέρα λοιπόν από την ερώτηση που έκανα στην Επιτροπή, θέλω να ρωτήσω και τον ε, εισηγητή. Η διάσκεψη αυτή πιστεύει μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτά που έχει γράψει ήδη στην έκθεσή του και πώς ε, τον κάνει να νιώθει αυτό που δήλωσε ο Πρόεδρος των 20 ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των πρώτων υλών και τις πρώτες ύλε τις ίδιες. Δηλαδή για το σιτάρι, ο συνολικός όγκος απολύεται 50 φορές χωρίς να αλλάζει η ιδιοκτησία για κερδοσκοπικούς λόγους και αν υπάρχει ένας οικονομικός παράγοντας που μπορεί να πληρώσει, μπορεί να αγοράσει 7% ε, του συνόλου της παραγωγής ε, κακάο, που είναι το 15% της συνολικής παραγωγής. Αυτή λοιπόν η έλλειψη σταθερότητας, η κερδοσκοπία δηλαδή, Εννοείται ότι φέρνει σε δύσκολη θέση τους αγρότες που δεν είναι κερδοσκόποι. Άρα η διαπίστωση αυτή μας κάνει πιστεύω να σκεφτούμε μήπως χρειάζεται μια ρύθμιση των αγορών των πρώτων υλών. Ο εισηγητής έχει γνώμη γι' αυτό και το κοινοβούλιο μας μήπως έχει χρέος να ξεκινήσει μια πολιτική συζήτηση με τα υπέρ και τα κατά δηλαδή. ώστε να δούμε τι γίνεται με την αγορά των παραγόγων στην αγορά πρώτων υλών και πώς εξελίσσεται η αγορά αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Este un raport... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπιουτικόφερ για την εξαιρετικά καλή αυτή έκθεσή του. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι στο μέλλον οι θέσεις εργασίας θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. Η ανταγωνιστικότητα δηλαδή στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. Εάν δηλαδή η Ευρώπη σε κάποιου τομεί δεν έχει πρόσβαση σε κάποιε πρώτε ύλε, η παραγωγή θα μεταφερθεί στους, στους τόπους όπου είναι διαθέσιμε αυτές οι πρώτες ύλες και έτσι ε, ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν εργαζόμενοι από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το τονίζει ο συνάδελφος Κόφερ στην έκθεσή του. Σε εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ή με κάποιες περιφέρειες, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και κεφάλαιο για τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. Ταυτόχρονα χρειάζονται επενδύσεις ε, για τις ε, τεχνολογίες ώστε να επιτρέψουμε μια αηφόρο ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Το 30% των αποβλήτων ουσιαστικά είναι δευτερεύοντα ε, προϊόντα τα οποία δεν ε, εκμεταλλευόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή στην στάση μας ως καταναλωτές. Χρειάζεται λοιπόν ε, να προσέξουμε περισσότερο αυτήν την έννοια του urban mining. Ε, την δυνατότητα δηλαδή ανακύκλωσης ε, ε, σπανίων γεών ή πολύτιμων μετάλλων. Να ξανασυγχαρώ τον κύριο Μπιτικόφερ, διότι είναι σημαντικό να καλέσουμε την Κομισιόν να δημιουργήσει νέες ε, στρατηγικές ε, για την ε, πρόσβαση στις σπάνιες γέες και στις πρώτες Όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος των σπανίων γεών, θα πρέπει να υπάρχει και στρατηγική πέρα από αυτόν τον απλό κατάλογο, ο οποίος να αντικατοπτρίζεται και στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όντω πολύ σύντομο. Και αυτό γιατί υπάρχει συμφωνία και είμαστε ευγνώμονε στον κύριο Μπουτικόφερ για την εξαίρετη, όπως είπαν και άλλοι ομιλητέ έκθεσή του. Είναι πολύ ισορροπημένη και πλήρης. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα-δύο σημεία μόνο έχω να θίξω. Δυστυχώς είναι εκεί όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας κάπως. Το ένα σημείο είναι αυτό που έχει να κάνει με υποστόχους, sub-targets. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και εμείς στις δικές μας προτάσεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες. Αλλά βρίσκουμε ότι είναι δύσκολο να βάλουμε νούμερα για τους σπόρους. Γιατί ο κίνδυνος είναι ότι είτε δεν θα είναι ρεαλιστικά τα νούμερα, είτε δεν θα έχουν επιστημονική βάση. Οπότε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να αγωνιστούμε για να το πετύχουμε κάποια στιγμή, αλλά πρώτα ας καθορίσουμε δείκτες ανά τομέα και μετά ας προσπαθήσουμε συνολικά να βάλουμε στόχους. Δεύτερον, έχει να κάνει με τη φορολόγηση. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Η ανησυχία μας είναι ότι σε σχέση με τις πρώτες ύλε. οι πρώτες ύλε χρησιμοποιούνται παντού στον κόσμο. Εφόσον λοιπόν επιβάλλουμε κάποια φορολόγηση στις πρώτες ύλε, αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι οι βιομηχανίες που τις χρησιμοποιούν θα βρίσκονται σε δυσμενή θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό παγκοσμίω. Αυτή είναι η συνέπεια. Βέβαια, και το έχουμε συζητήσει και με το Κοινοβούλιο, υπάρχουν ενδεχομένω και άλλοι τρόποι. Αν βρούμε λοιπόν τρόπο να αντικαταστήσουμε ένα είδος φορολόγησης από κάποια άλλη, από κάποιο άλλο είδος, τότε ίσως να είναι αλλιώ τα πράγματα και να συμφέρει. Αλλά χρειάζεται να αναλυθεί σε βάθο το θέμα πρώτα. Τέλος, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, η ιεράρχηση των πρώτων υλών. Αναφερθήκατε στην ιεράρχηση των αποβλήτων, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, σαν ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί βλέπετε χρειάζεται ανάλυση ολόκληρου του κύκλου ζωής και το αναγνωρίζουν όλοι αυτό ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια ανάλυση. Δεν χρειάζεται να μπω τώρα σε λεπτομέρειες και σε παραδείγματα. Η αξιολόγηση πάντως αυτή, ολόκληρου του κύκλου ζωής, είναι ζωτική σημασία. Και τώρα το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πολλά από τα θέματα που θίξατε και είδα, είπατε για τη διάσκεψη τη χθεσινή της Κομισιόν, τη Κομισιόν, το Συμβούλιο να γνωρίζουν ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε νομοθεσία όταν προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ρύθμιση στην ανακύκλωση. Αλλά αν δεν είμαστε σε θέση να καινοτομήσουμε είτε μέσω της τεχνολογίας, είτε μέσω άλλων πιο στάνταρτ ιδεών, αν δεν θίξουμε τέτοια ζητήματα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τα επόμενα δέκα χρόνια να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με μια έκκληση. Κατά σύμπτωση, υπάρχει μια διαβούλευση στο διαδίκτυο για την ιδέα καινοτομίας ε, όσον αφορά την κατανομή των πρώτων υλών. Είναι μια ευκαιρία και γι' αυτό θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των Ευρωβουλευτών. Ίσως τις εκλογικές σας περιφέρειες να θέλουν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Και να, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, να εκφράσω τις ε, ευχαριστίες μου. Ο κύριος Σεσιμάνσκι είχε δίκιο πριν που είπε ότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας έχει βελτιωθεί με τις ε, τροπολογίες. Και ήταν πολύτιμες και οι προτάσεις που ακούσαμε σήμερα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να τις σχολιάσω. Να ξεκινήσω από το ερώτημα της κυρίας Δελκαστήγιο σχετικά με τη συμβαστική τροπολογία 4. Το κείμενο αυτό το εκπονήσαμε για να λάβουμε υπόψη μας την επιθυμία και των συναδέρφων ε, να έχουμε ευρύτερη οπτική. Το είπε αυτό και η κυρία Ουλφσκοκ. Δεν νομίζω ότι θα αποτύχουμε με τη συγκεκριμένη διατύπωση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα. Είμαι αισιόδοξο. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι τόνισαν τη θέση ότι δεν ε, χρειάζεται να συζητάμε εδώ για την κάθε πρώτη ύλη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια σημεία, διότι αλλιώς θα χάσουμε τελείως τον έλεγχο. Πάντως ε, νομίζω ότι σχετικά με αυτή την πολιτική θέση που εκφράσατε, νομίζω ότι μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά την παρατήρηση της κυρίας Χολ, Και όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, συμφωνώ με όλα όσα είπατε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, πετύχουμε και την έγκριση της πλειοψηφίας. Να επανέλθω στο ερώτημα της κυρίας ε, Ουλφ Σκόκ και της κυρίας Μερκής. Τι φωτογραφίζουμε εδώ, τι λαμβάνουμε υπόψη μας, ε, σε στρατηγικές για την αποτελεσματικότητα, σε ε, διάφορα μέσα όσον αφορά την ε, διπλωματία των πρώτων υλών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ούτως ή άλλως ισχύουν και για τις διάφορες πρώτες ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύτιμο το θέμα αυτό. Ο κύριος Σιμάνσκι ανέφερε ότι υπάρχουν διάφορες στάσεις ε, για να προταθούν ε, ε, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Και είπε ότι αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει μετά από μελέτη αντικτύπου ώστε να αποφύγουμε ε, να ε, έχουμε πλεόνασμα νομοθετικών ρυθμίσεων όσον αφορά τους συγκεκριμένους στόχους. Πρέπει να ομολογήσω ότι ε, τώρα πια είμαι λιγότερο τολμηρός από ότι ήμουν στην αρχική πρόταση όπου είχα συμπεριλάβει συγκεκριμένο μετρήσιμο στόχο διότι Θέλουμε να πετύχουμε συνένεση και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλύτερη, πιο έξυπνη προσέγγιση η συγκεκριμένη. Ε, εάν υπάρχουν παράμετροι για, τη, για τον υπολογισμό των στόχων, τότε νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να θέσει τους στόχους αυτούς και όχι η και όχι το κοινοβούλιο. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Τζαβέλα για τον ε, έλεγχο και τη ρύθμιση του εμπορίου, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν κατάλαβα ακριβώ τι εννοείται. Θα παρακαλούσα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό διμερώς μετά. Είμαι κάπως ε, προσεκτικός, επιφυλακτικός όσον αφορά την ιεράρχηση των πρώτων υλών. Τίνω προς την κατεύθυνση του κυρίου Τεκαβάλιο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε μια τέτοια ιεραρχία. Εάν θέλουμε μια τέτοια ιεραρχία, πόσο κατευθυντικοί θα είμαστε. Νομίζω ότι μέσα της αγοράς ε, είναι καλύτερα για να ε, δοθούν τέτοιες κατευθύνσεις. Παρά η πολιτική. Εφόσον βέβαια έχουν καθοριστεί σωστά οι οικολογικές ε, προϋποθέσεις πλαισίου. Επίσης, όσον αφορά την ε, παρατήρηση ότι ε, η ενεργειακή αξία θα αποτελεί μέτρο, μπορεί αυτό να είναι ένα μέτρο, όχι όμως το μοναδικό. Αυτό που είπε ο κύριος Κίπερ, δηλαδή. δεν μπορούμε όλα να τα ε, ε, εξετάζουμε υπό το φως ενεργειακής αξίας και όσον αφορά το θέμα ε, των φόρων που αναφέρατε η κυρία Κύριε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δηλαδή ε, αντικατάσταση των φόρων, όχι αύξηση. Αλλά είμαι αρκετά επιφυλακτικό στο θέμα αυτό και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Καταρχήν, εάν ο τόνος ε, χαλκού στοιχίζει 10.000 ευρώ, τότε αναρωτιέμαι πόσο υψηλός θα πρέπει να είναι ο φόρος ε, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε την αγορά. Τη στιγμή που είναι τόσο υψηλές οι τιμές, ε, αμφιβάλλω αν οι φόροι μπορούν να έχουν κάποια επίπτωση. Και επίσης θα πρέπει να είναι τόσο διαφοροποιημένοι οι φόροι αυτοί που μπορεί να καταλήξουμε σε λανθασμένη κατανομή. Δηλαδή να επενδύσει κανείς σε κάποια πρώτη ύλη επειδή αξίζει τον κόπο από πλευράς φόρων παρότι ε, οικονομικά κατά τα άλλα δεν έχει κανένα νόημα μια τέτοια επένδυση. Και τέλος ε, το θέμα είναι πόσο γραφειοκρατικό θα είναι τέτοιο σύστημα Ε, εάν θέλουμε να ε, ε, συμπεριλάβουμε 17 τέτοιε σπάνιε για σε ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είμαι κατά μια τέτοια πρόταση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όσον, αφορετε, όσον αφορά τι παρατηρήσει του. του κυρίου Σκάλας, νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει ε, από μόνη της ε, να ορθοποδήσει, αλλά Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τις σπάνιες γεές, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και θέμα ε, διαθεσιμότητας ε, των απαραίτητων δεξιοτήτων, αλλά και των και των σταδίων επεξεργασίας. Η Κίνα δεν έχει μόνο τη μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά έχει ε, και σχεδόν αποκλειστικότητα όσον αφορά τα τρία πρώτα στάδια επεξεργασίας των σπανίων γεών. Τίθενται λοιπόν πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές πολιτικές αντιθέσεις, διότι εν μέρη στο Κογκρέσο προτάθηκε να γίνεται η επεξεργασία εντό των Ηνωμένων Πολιτειών και να ε, δοθούν δάνεια για κάτι τέτοιο, ενώ ε, άλλο μέρος του Κογκρέσου ε, ήταν κατά κάτι, εναντίον αυτού. Όσον αφορά το να υπάρχει ένα σχέδιο μέχρι το 2050, νομίζω ότι έχω συμπεριλάβει σχετική διατύπωση. Νομίζω όμως ότι όπως πρότεινε η Κομισιόν, νομίζω ότι θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να εξετάζουμε ποιες πρωτεσίλες είναι οι κρίσιμες ανα πάσα στιγμή. Διότι αυτό μπορεί να αλλάζει από εποχή σε εποχή. Όσον αφορά ε, την ε, αποθεματοποίηση, το stockpiling, ε, είμαι αρκετά επιφυλακτικός. Έχω συζητήσει με αρκετούς άκουσα κάποια πιστικά ε, ε, ε, επιχειρήματα, αλλά πώς μπορώ να δημιουργήσω αποθέματα τη στιγμή που δεν έχω καλά-καλά να καλύψω τις καθημερινές μου ανάγκες. Για κάποιες πρώτες πάντως σίγουρα έχει νόημα και διαπιστώνω ότι στην Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών υπάρχει προσπάθεια ε, τουλάχιστον ε, να καταλήξουν σε κοινέ ε, στρατηγικές αγοράς πρώτων υλών. Εάν η βιομηχανία δεν είναι καν σε θέση να συνεργαστεί για τέτοιους τομείς, τότε είναι αμφίβολο αν το κράτος είναι σε θέση να δημιουργήσει αποθέματα τέτοιων πόρων. Ο κύριος Οντί ε, ε, ρώτησε σχετικά με την εχθεσινή διάσκεψη. Κύριε Οντί, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Προσπάθησα να δω αν ήταν δυνατόν ε, να συμμετάσχω εκεί. Μου είπαν ότι προβλέπονταν... τόσοι σπουδαίοι ομιλητές, ε, περίμενα τόσους σπουδαίους ομιλητές ε, εκ των οποίων το, ε, ε, υπήρχε μεγάλο ποσοστό Γάλλων. Ε, μου είπαν λοιπόν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να συμμετάσχει και κάποιος ευρωβουλευτής. Αλλά εγώ συνέβαλα στο newsletter, στην, στο ενημερωτικό φυλάδιο που δημοσιεύτηκε σχετικά με αυτήν την διάσκεψη. Η διάσκεψη ε, αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ε, πίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Η ΕΚΟΝ ε, είπε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα, γιατί έχουμε τώρα πάρα πολλή δουλειά. Θα επανέλθουμε στα πλαίσια της οδηγίας MIFID. Είναι αυτό το λεγόμενο financialization of commodities. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το, με το οποίο θα ξανασχοληθούμε στα πλαίσια της οδηγίας MIFID. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν τώρα να έχουμε επικάλυψη των σχετικών εργασιών. Ε, δύο σημεία έχω ακόμα, λέει ο μιλητής. Η κυρία Τίκα Αναφέρθηκε στην ε, μεταφορά σε τρίτες χώρες ε, της ε, παραγωγής. Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί το ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η μεταφορά αλλού της παραγωγής δεν είναι καν δυνατότητα και ότι έτσι θα εξαφανιστούν τελείως. Και επίσης συμφωνώ με την παρατήρηση που έγινε. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν να ξεπεράσουν την αντίσταση του ενός κράτους μέλους που έχει μπλοκάρει αυτήν την κατά άλλα πολύ καλή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κύριε Σοντή. Euh, πολύ σύντομα. Δεν πρόκειται για την εσωτερική γαλλική πολιτική. Πρόκειται για την ομάδα των 20. Προσθέτω, όπω και όλη παρατήρηση που έκανα σήμερα το πρωί και τώρα, λέω, να προτείνετε στην Επιτροπή, μάλλον να διαμαρτυρηθείτε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι σκανδαλώδε να μην προσκαλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια διάσκεψη που οργανώνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιου επίπεδου. Ενώ έχουμε το θέμα αυτό, έχουμε συγητή, αποφασίζουμε για αυτό το θέμα και δεν μας ζητάνε να συμμετέχουμε για να αξιολογήσουμε καλύτερα. Και επιπλέον μαθαίνω ότι ο υπεύθυνο εισηγητής ήθελε να πάει και του αρνήθηκα την πρόσβαση. Προτείνω λοιπόν να διαμαρτυρηθούμε επίσημα. Τέλος, <clears throat> συνάδελφοι. Λέτε 22% Γάλλοι. Μα ξέρετε ότι η ομάδα των 20 δεν έχει διοίκηση. Οπότε αυτός που προεδρεύει έρχεται, όπως και η Ουγγρική Προεδρία, έρχεται με τους Ούγγρους υπαλλήλους της. Οπότε Πρόεδρε, το μόνο που προτείνω είναι μία επίσημη διαμαρτυρία. Τίποτα άλλο. Εάν ήταν εκδήλωση της ε, Κομισιόν, τότε σαφώς θα ε, διαμαρτυρηθούμε πολύ σοβαρά. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι ε, μας εμπόδιζαν να παρακολουθήσουμε, αλλά μας εμπόδισαν την ενεργό συμμετοχή. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δεν δεν μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε ενεργά. Ωραία, ε, έτσι κλείνουμε το θέμα αυτό της ημερήσιας ε, διάταξης. 30 Ιουνίου έχουμε την ψηφοφορία. Κλείνω τη συνεδρίαση και σε δύο λεπτά θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ οι άλλοι συνάδελφοι, οι προσκεκλημένοι, να εγκαταλείψουν γρήγορα την αίθουσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ.